Public hearing on IFRS 9. Καλησπέρα σας. Μπορούμε να ξεκινήσουμε την δημόσια μας ακρόαση για το ε, χρηματοπιστωτικό μέσο που όπως ξέρετε θα πρέπει να αντικαταστήσει το ε, ισχύον και θα αρχίσει να ισχύει από την 1η 2018. Με τη νομική διαδικασία που θα έχει ολοκληρωθεί, ήδη κάναμε την ε, έγκριση των συμβουλών με τη συμβουλευτική ομάδα ΕΦΡΑΓ. Παρακολουθήσαμε στενά όλες τις εξελίξεις για αυτό το θέμα και Είχαμε ήδη τρεις συνεδριάσεις όπου το συζητήσαμε με εκπροσώπους της ΕΦΡΑΚΑ και της ΙΤΙΝΙΑΣΠ, την... Ε, τα διεθνή πρότυπα και τώρα θα συζητήσουμε το θέμα με τέσσερις σημαντικούς εμπειρογνώμονες, τους οποίους και θέλω να ευχαριστήσω που είναι σήμερα ε, εδώ ή στη Washington, εν πάση περιπτώσει, online. Αντρέας Βακρόου, που είναι πρόεδρος της Επιτροπής ε, προτύπων, Λογιστικών Προτύπων της Γερμανίας, τον Νικολάς Βερόν, από το Ινστιτούτο Πέτερσον, τον Ανδρέας Χάκερ, από την ε, Συνεταιριστική Τράπεζα Γερμανίας και τον Μάικλ Χάσλεϊ, πρόεδρο της ΕΦΡΑ ΤΕΚ και πρόεδρο της ε, Ομάδας Εργασίας για τα χρηματοπιστωτικά μέσα. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε όλοι εδώ. Θα συζητήσουμε διάφορα συγκεκριμένα ζητήματα, όχι μόνο γενικά για το IFRS 9, Καταλαβαίνω πως υπάρχει ένα σημαντικό σημείο που αφορά τις ασφαλίσεις και την αναντιστοιχία τους με το IFRS 4, καθώς και τις διάφορες επιλογές που είναι υποσυζήτηση και διάφορα άλλα σημαντικά σημεία, τα οποία θα συζητήσουν οι πυρογνώμονές μας με τους οποίους και θα ξεκινήσουμε. Έχετε πέντε λεπτά έκαστος και ο πρώτος ομιλητής είναι ο Ανδρέας Μπάκρο. Έχετε το λόγο. Πρόεδρε Γκουαλτιέρη, κυρίες και κύριοι, σας ε, είμαι ευγνώμη που δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω σήμερα για το IFRS 9, το οποίο εξεδόθη το 2014, ύστερα από έξι χρόνια εκταμένων συζητήσεων με τους βασικούς ε, ενδιαφερόμενους φορείς. Έξι χρόνια φαίνεται να είναι μακρύς χρόνος για την ανταπόκριση στην χρηματοπιστωτική κρίση, ωστόσο τα προϊόντα και οι αγορές ε, συνεχώς αλλάζουν, οι κανονισμοί, η εποπτεία εξαρτώνται περισσότερο από τα λογιστικά στοιχεία από ό,τι παλιότερα και ε, τα στοιχεία αυτά αλλάζουν επίσης. Το πακέτο IFRS 9 ανταποκρίνεται σε αυτές τις προκλήσεις ε, και στα χρηματοπιστωτικά ε, μέσα και αφορά τους ομίλους, παραγωγούς, μεταποιητές και παρόχους υπηρεσιών. Αυτές οι υπηρεσίες προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν παραδοσιακά μη δομημένα προϊόντα όπως ε, τα δεκτά ε, και τα, και παράγωγα ο πρόεδρος διακόπτει και ζητά από τον ομιλητή να μιλήσει λίγο πιο αργά, γιατί διαφορετικά οι διερμηνείς δεν μπορούν να σας ακολουθήσουν, να σας παρακολουθήσουν. Apologies. Some entities may engage. Ορισμένες, ορισμένοι όμιλοι καταφεύγουν σε παράγωγα ώστε να εξασφαλίσουν ε, την ασφάλειά τους απέναντι στους, ε, στις κειμενόμενες διεθνείς τιμές των διαφόρων αγαθών. Για αυτούς όμως το FRS 9 θα βελτιώσει ε, τις αναφορές τους και την καταγραφή των λογιστικών τους, ε, συμβάλλοντας έτσι στην διαφάνεια. Σε όλους τους άλλους τομείς, στις ε, ακραίες περιπτώσεις, οι όμιλοι θα, χρησι... θα να συνεχίσουν να καταγράφουν τα χρηματοπιστωτικά τους μέσα με το δικό τους τρόπο, το γνωστό τρόπο, και έτσι οι στρεβλώσει θα ε, ελαχιστοποιηθούν. Αστραφώ τα χρηματοπιστωτικά Ινστιτούτα και ιδιαίτερα τι τράπεζες. Υπάρχουν δύο βασικοί τομεί όπου το IFRS θα αλλάξει τον τρόπο λογιστική των τραπεζών λόγω τη χρηματοπιστωτική κρίση. Καταρχήν, οι νέε απαιτήσει για την κατανομή των χρηματοπιστωτικών μέσων ανάλογα με το επιχειρηματικό του μοντέλο σημαίνει πω οι όμιλοι αυτοί δεν θα μπορούν πλέον να καταγράφουν τα μη παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά μέσα στο κόστο του και να κρύβουν έτσι τον κίνδυνο που εμπεριέχεται σε αυτά τα μέσα. Γι' αυτό και η μεγάλη ερησιμότητα αλλά και η μόχλευση θα πρέπει να αναφέρονται και έτσι θα είναι ορατός οποιοδήποτε αντίκτυπος ε, αλλαγών ή κινδύνου και θα συμβάλλουμε έτσι στην διαφάνεια. Τώρα, Μπορεί κανείς να διερωτηθεί κατά το πόσο το IASB έχει βρει τη σωστή διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στα διαρθρωμένα, τα δομημένα και τα μη δομημένα προϊόντα, αλλά βασικά πιστεύω πως η προσέγγιση αυτή είναι η λογική. Κατά δεύτερο λόγο, το σε e νέα συμπεριλαμβάνει ένα τελείως νέο πρότυπο, ε, το οποίο θέλει να διατηρήσει την ε, εικόνα, μια μακροχρόνια εικόνα της απόδοσης κάποιας ε, τράπεζας. Η ανάπτυξη αυτών το, του μοντέλου ε, της αναμενόμενης απώλειας ε, πιστοληπτικής ικανότητας είναι αυτό το οποίο θα καταστήσει περισσότερο διαφανή την κατάσταση. Κάποιος πελάτης είτε αποδίδει είτε όχι. αλλά δεν είχαμε μέχρι τώρα αρκετά στοιχεία ώστε να μπορούμε να συνδυάζουμε αυτά τα δύο σημεία χρονικά και δεν υπήρχαν ενδείξεις για το τι δεν πήγαινε καλά. Τώρα, κατα... το... οι αλλαγέ στην πιστοληπτική ικανότητα οποιοδήποτε ομίλου ή τράπεζα θα γίνεται εμφανή ε, γρηγορότερο λόγω τη καταγραφή της ε, απόδοση ή τη μη απόδοσης ε, της τράπεζας. Και αυτή είναι μια σημαντική βελτίωση. Τώρα για την, ε, τις ασφαλιστικές Ενώ πολλά από τα επιχειρήματα που, γίνονται τις, που σας ανέφερα για τι τράπεζες συνισχύουν και για τι ασφαλιστικέ εταιρείε, υπάρχει μια σημαντική διαφορά. Γιατί βασικά ε, καταγράφουν εκείνες ε, τις ε, το παθητικό τους στα ισοζύγια τους, στους ισολογισμούς τους, ε, με συγχωρείτε. Όμως αυτό γίνεται όταν δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί η κατάσταση και θα υπάρχει διαφορετική επίπτωση από ότι στο IFRS 4. Στο IFRS 9 έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό το πρόβλημα, το οποίο οφείλεται στις διαφορετικές ημερομηνίες. Ελπίζουμε πως η Ευρώπη θα βαρύνει με το κύρος της αυτή τη συζήτηση και θα συνεργαστεί για την εξέβρεση μιας διεθνούς λύσης. Διαφορετικά θα εγκριθεί ίσως ή θα υπάρχει κάποια αλλαγή, ότι θα έχει ισχύσει το IFRS 9 για κάποια χρόνια στην Ευρώπη. Θα ολοκληρώσω λέγοντας ότι ποτέ δεν πρόκειται να βρεθεί τέλεια λύση. Θα πρέπει βήμα-βήμα να προχωρήσουμε και ως προς αυτό πιστεύω πως το IFRS 9 αποτελεί ένα καλό και προφανές καλό βήμα, θετικό βήμα προς μια διαφανέστερη κατάσταση και έτσι θα διευκολύνει και την Ευρώπη να συμβαδίσει με τον υπόλοιπο κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε και με τα χαρά θα απαντήσω σε οποιαδήποτε, οποιαδήποτε ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής από τη Washington, ο Νικόλας Βερόν. Δεν ξέρω αν με ακούτε. <clears throat> Σας ακούμε. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ ε, που με καλέσατε σε αυτή την ακρόαση και θα ήθελα να ευχαριστώ κυρίως ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ότι επιθυμεί και θέλησε να καταθέσω μέσω τηλεδιάσκεψης κάτι για το οποίο ευθύς εξ αρχής ε, ζητώ συγγνώμη αλλά επειδή δεν είχα άλλη δυνατότητα δεν μπορούσα και να τα αποφύγω. Σε μεγάλο βαθμό συμφωνώ με αυτά που ελέγχθησαν επί του τεχνικού αλλά θα ήθελα να προσθέσω ορισμένα πράγματα όσον αφορά την governance που νομίζω ότι είναι κάτι που εξετάζει για πρώτη φορά η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το IFRS 9. Το IFRS 9, το εργαλείο αυτό, ταυτίζεται με την ουσία αυτών που ελέγχθησαν η G20 στο Λονδίνο, όπου αποφασίστηκε να περάσουμε σε ένα άλλο μοντέλο Άρα δηλαδή κατά κάποιον τρόπο υλοποιείται αυτή η επιθυμία με έναν σωστό τεχνικό τρόπο. Η προσέγγιση επικρίθηκε γιατί διαφέρει από την πρόταση ε, του Συμβουλίου EFSB των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά νομίζω ότι περισσότεροι παρατηρητές και εμπειρογνώμονες συμφωνούν ότι η προσέγγιση του Οργανισμού Διεθνών Λογιστικών Προτύπων ISB ε, είναι ε, σωστή ε, και δεν υπάρχει κανένας λόγος ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδιώξει την ταύτιση των κοινοτικών με τα διεθνή πρότυπα. Υπάρχουν λόγοι γιατί τα δύο αυτά πρότυπα δεν συγκλίνουν. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να συζητηθεί κυρίως στις Ηνωμένε Πολιτείες. Ε, δεν νομίζω ότι είναι κάτι ε, που θα μπορούσε να κρατήσει όμοιρο το χρηματοψηφικό εργαλείο υπαριθμών 9. Υπάρχουν και κάποιες ε, αντιρρήσεις για το εργαλείο αυτό από μια μικρή ομάδα επενδυτών, επαγγελματιών του κλάδου και από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι εστιάζουν στο κατά πόσον είναι θεμητή όλη αυτή η άποψη. Υπήρχε κάποια αντιπαράθεση για μεγάλο κονικό διάστημα στηριζόμενοι και με νομικά επιχειρήματα. Κατά την άποψή μου όμως αυτοί δεν μπαίνουν στην ουσία του εργαλείου αυτού, ε, δεν επηρεάζονται οι Ευρωπαίοι επενδυτές και για το λόγο αυτό τα επιχειρήματα που προβλήθηκαν δεν θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την έγκριση του εργαλείου IFRS 9. Και αναφέρομαι εδώ κυρίως σε αυτά που λέξαν από οργανισμούς όπως είναι ε, τοπικά συνταξιωτικά εργαλεία ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο και αλλού. Ο προηγούμενος ομιλητής τοποθετήθηκε. Εγώ νομίζω ότι οι ε, επιφυλάξεις που έχουν σχέση με τις ασφάλειες πρέπει να ληφθούν υπόψη, όμως να το πω κάπως αλλιώς. Οι επιφυλάξεις αυτές <clears throat> θα αντιμετωπιστούν κατά πάσα πιθανότητα από τον οργανισμό ISB ξεχωριστά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 θα ε, διαπιστωθεί, θα διαπιστωθούν οι επιπτώσεις ε, του εργαλείου αυτού από το ISB, αλλά όλα αυτά δεν είναι καθοριστική σημασία από την πλευρά της αγοράς και της ασφάλειας όπως το παρουσιάζουν κάποιοι ασφαλιστές. Και δεν πρέπει αυτές οι επιφυλάξεις να αποτελούν προϋπόθεση για την έγκριση του IFRS 9. Να αναφερθώ τώρα λιγάκι και στην γραπτή μου εισήγηση. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει ουσιαστικά στη συνεχιζόμενη επιτυχία του εργαλείου IFRS. Ε, δεν μπορώ να σκεφτώ κανένα άλλο εργαλείο με τη μορφή διεθνών χρηματοψηφιακών προτύπων όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση να ήταν πιο επιτυχημένη. Και εννοώ ότι επειδή ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το εργαλείο πριν από 10 χρόνια, γι' αυτό διαδόθηκε το εργαλείο αυτό και κατέληξε σε μεγάλη επιτυχία, επιβάλλεται σε όλο τον κόσμο ε, και αναστέλει αρνητικές επιπτώσεις. Αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός στρατηγικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα πρέπει να συμφωνεί σε όλα όσα προτείνει ο οργανισμός ISB. Υπάρχουν ε, κάποια εργαλεία και κάποιοι τομείς ε, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως έχει σημειώσει επιτυχία σχετικά πάντα με το IFRS. Υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις ως προς το governance, την διαχείριση των προτύπων του IFRS που συντάσσονται από το ISB. Όλα αυτά ε, θα συνεχίσουν να συζητούνται. Σε αυτή τη στιγμή είναι σε πειραματική φάση, τίποτα δεν έχει ολοκληρωθεί, χρήζουν βελτιώσεων, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που πρέπει να βελτιωθούν, αλλά είναι σωστή η συζήτηση που γίνεται. Εγώ σχετικά με τη διαχείριση πιστεύω ότι η συζήτηση αυτή θα πρέπει να είναι ξεχωριστή από τα ε, εσωτερικά πρότυπα, γιατί αλλιώς θα υπάρξει ζημιά ε, κυρίως για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ασκεί επιρροή στον καθορισμό του IFRS 9. Είναι ένα θέμα που έχει σχέση με το να μπορέσει κανείς να συνδυάσει την έγκριση του εργαλείου και την ε, σωστή εποπτεία, κάτι το οποίο γίνεται τώρα από ξεχωριστούς οργανισμούς όπως είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Εθνικές Αρχές και την ΕΣΜΑ. Και τέλος, για να ολοκληρώσω, ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι του θεματοφύλακα σε αυτή τη διαδικασία. Κατ' ουσίαν θα έπρεπε το Κοινοβούλιο να πει όχι στην έγκριση του εργαλείου αν είχαν αποτύχει τα πάντα και να έπρεπε το Κοινοβούλιο να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των πολιτών. Ε, πριν από λίγα χρόνια συνέστηνα ε, να απορρίψει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το προηγούμενο εργαλείο το οποίο κατά την άποψή μου δεν εξυπηρετούσε τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Εγώ δεν είμαι υπεραμήντορα στη ASB, αλλά στην περίπτωση αυτού του εργαλείου του ΕΝΕΑ είναι σαφές ότι τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προστατεύονται παρκώς από μια κανονική διαδικασία και από αυτά που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που θα συνεχίσει να κάνει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει κανένα λόγο να καταθέσει βέτο ε, ο έλεγχος, βεβαίως ο εντελεχής έλεγχος που κάνει κάθε φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σωστός και θεμητός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Ανδρέας Χάκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δώσατε να λάβω το λόγο και θα ήθελα με αυτήν την ευκαιρία να σας παρουσιάσω λιγάκι και την άποψη των ε, γερμανικών συνεταιρισμών, γενικότερα την άποψη ε, ε, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εμείς έχουμε περίπου 20 εκατομμύρια μέλη και ε, έχουμε πάρα πολλές συνεταιριστικές τράπεζες οι οποίες δεν χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο αλλά το απορρίπτουν κατηγορηματικά. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο εγώ έχω μια λιγάκι διαφορετική άποψη όσον αφορά το εργαλείο IFRS από ότι ο Γερμανός νομοθέτης ε, και πρέπει να σας πω ότι δεν εκπλήσωμαι που δεν <clears throat> αντιμετωπίζει το εργαλείο αυτό ως ε, ιερό και άγιο και θα σας εξηγήσω τους λόγους γιατί τα πιστεύω όλα αυτά. Καταρχήν όσον αφορά το εργαλείο αυτό και συμφωνούν όλοι από αυτού είναι ένα σημαντικό εργαλείο της, ε, του χρηματοπιστωτικού τομέα. Νομίζω <clears throat> όλοι συμφωνούν από αυτού. Αν δει κανεί ποια είναι τα προβλήματα τα νομοθετικά αυτό το εργαλείο είναι καθοριστικής σημασίας για τα συμφέροντα και των μάνατζερ και των επενδυτών. Άρα δηλαδή εδώ ελοχεύει ένας σημαντικός κινδύνος και το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι οι ισολογισμοί. Πάμε στο EFRS 9. Κατά την άποψή μου αυτό δεν βελτιώθηκε σε σχέση με το 39 και στη τελική ανάλυση το περίφημο fair value οδήγησε σε μειοπική στάση. Η σταθερότητα μάλιστα του χρηματοπιστωτικού συστήματος υπονομεύτηκε. Γι' αυτό δεν με εκπλήττει το γεγονός ότι κάποια ασφαλιστικά ταμεία έχουν επιφυλάξεις. Το EFRS 9 θα αντικαταστήσει πλήρως το 39. Κατόπιν τούτου πρέπει να διερωτηθούμε ποιες είναι οι βελτιώσεις που θα προκύψουν, ε, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις ε, στον χρηματοψηφικό τομέα ως προς την ανάληψη κινδύνου και κατά πόσον μπορεί να εφαρμοστεί αυτό το εργαλείο. Έχουμε δύο τομείς. Ο ένας αφορά το fair value και τους ισολογισμούς και ο δεύτερος τομέας ε, αφορά το κόστος εφοδιασμού. Θα περιοριστώ στο πρώτο. Το fair value, η θεμητή τιμή, δεν είναι απλά η τιμή αγοράς. Είναι μια τιμή η οποία προκύπτει καθαρά θεωρητικά. Δηλαδή, σε περίπτωση εμφιβολίας, σας λέω, είναι καθαρά θεωρητική τιμή και δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την πραγματική τιμή της αγοράς. Όμως οι, ε, ε, τα λογιστικά πρότυπα χρησιμοποιούνται παραδοσιακά για την ενημέρωση των αγορών. Τώρα λοιπόν ενημερώνουμε τις αγορές εγγράφοντας αυτήν την αξία στους ισολογισμούς. Στην καλύτερη λοιπόν των περιπτώσεων ε, αυτό είναι άχρηστο. Στη χειρότερη των περιπτώσεων μιλάμε για ένα εργαλείο προκυκλικό το οποίο οξύνει περαιτέρω της κρίσεις. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι αυτή η fair value, αυτή η θεμητή αξία δίνει στοιχεία ε, στους ισολογισμούς που είναι υψηλότερα από τα παραδοσιακά. Δηλαδή ε, είναι πιο ε, δαπανηρή η απόσβεση και είναι πολύ πιο εύκολο οι σχετικές αξίες να εκτιναχτούν στα ύψη. Το εργαλείο αυτό, το υπαριθμόν 9, δεν επέφερε καμία βελτίωση και αυτό δεν μας εκπλήσει, γιατί πρέπει κανείς να διορτηθεί τι κρύβεται από πίσω. Τα λογιστικά πρότυπα από τον νομοθέτη ε, ανατέθηκαν σε ιδιώτες, δηλαδή τα λογιστικά πρότυπα διεθνοποιήθηκαν, καλό είναι αυτό, αλλά προέκυψε και με τον τρόπο αυτό ένα μονοπόλιο. Και τα λογιστικά πρότυπα συγκεντρώθηκαν σε μία και μόνο βάση, άρα δηλαδή, όπως ανέφερα σε μία μελέτη μου, ε, την οποία είχα προετοιμάσει εν ώψη της συνεδρίασής μας, όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την αγορά. Η σύνθεση του Οργανισμού Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, του ESB, κατ' ουσίαν ε, ήταν αυτό που περίμενε κανείς και ε, σε σχέση με το εργαλείο. Δεν προκύπτει καμία χρησιμότητα. Η εποπτεία χρειάζεται μια ενιαία βάση, άρα δηλαδή θα πρέπει κανείς να είναι σαφής και να γνωρίζει ότι η σύγκληση μόνη της και η εφαρμογή σε παγκόσμιο επίπεδο δεν επιφέρουν από μόνα τους βελτίωση, γιατί αν ε, η οικονομική κατάσταση είναι αρνητική, το ίδιο ισχύει και για τα ε, αργαλεία που χρησιμοποιούνται για τους ε, ισολογισμούς. Και σε τελική ανάλυση τι εξυπηρετεί αν όλοι συντάσσουν προκυκλικούς ισολογισμούς. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι το ESB δεν έχει τελικά δημοκρατικό έλεγχο. Δηλαδή οι κανονισμοί ε, δημοσιεύονται από εμπειρογνώμονες χωρίς να υπάρχει καμία σχέση με ερετά όργανα και στο τέλος κατατίθεται μία ολόκληρη δέσμη μέτρων. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να πει ή θα δεχθεί το σύνολο των μέτρων, όλη τη δέσμη ή τίποτα. Αυτό όμως δεν είναι δυνατόν, γιατί κατ' ουσία μπορεί κανείς να απορρίψει ένα πρότυπο ή η Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσει κάποια στοιχεία ενός προτύπου. Σε τελική ανάλυση υπάρχει ο σχετικός κανονισμός και θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι τα ε, μοντέλα που αφορούν ε, τις ε, μετρητές ε, συναλλαγές, τα μοντέλα αυτά δεν οδήγησαν απαραίτητα σε ασφάλεια και ασφαλή εφαρμογή των κανονισμών. Αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ πολύ. Και... Σας, ευχαριστώ. πολύ. Ο Μάικ Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας ε, κάνω μια εισήγηση σήμερα έχουμε να κάνουμε με διάφορες ε, παρεξηγήσεις ε, που νομίζω ότι έχουν γίνει σε σχέση με τα πρότυπα που προτείνουμε. Γιατί θα πρέπει να εγκριθεί το IFRS ε, 9, γιατί είναι μια βελτίωση όσον αφορά τις χρηματοπιστικές αναφορές, γιατί ανταποκρίνεται στο εξαιρετικά, στο, στην επίκριση που έλεγε ότι μέχρι τώρα συλλάγαμε πολύ λίγα και πολύ αργά στοιχεία είναι μια λογική συμβιβαστική λύση δεδομένων των πρακτικών εμποδίων που μπορεί να έχουμε. Δεύτερον, η αναγνώριση και η μέτρηση των χρηματοπιστωτικών μέσων βασίζεται περισσότερο στι αρχέ, στη δομή και στη συνοχή του και άρα δίνει περισσότερε σχετικέ πληροφορίε. Τρίτον, το λογιστικό μοντέλο είναι απλούστερο και πιο συμμορφωμένο προ τι επιχειρηματικέ πρακτικέ. Έχει αξιολογηθεί ότι συμβάλλει θετικά στην χρηματοπιστωτική σταθερότητα από την ECB και από την EBA, την Ευρωπαϊκή ε, Τραπεζική Αρχή. Ε, υπάρχει συνένεση υπέρ της έγκρισης σε σχέση με τα σώματα τα οποία σας ανέφερα προηγουμένως, τους οργανισμούς που ανέφερα, όπως η ΕΙΟΠΑ που προετοιμάζει ορκωτούς λογιστές και που προτείνει να εφαρμοστεί χωρίς απεραιτέρω καθυστέρηση. Η μη δευθυγράμμαση με, την, ε, με το στάνταρ της πραγματική ημερομηνία, αν και είναι μεταβατικό ε, θέμα, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζεται. Εν γέννη λοιπόν το IFRS 9 αναμένεται να εξυπηρετήσει τον κεντρικό στόχο του κανονισμού, δηλαδή υψηλή ποιότητα, διαφάνεια και συγκρίσιμες ε, αναφορές που είναι απαραίτητε για να στηριχθεί η ε, αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα της χρηματοπιστωτικής αγοράς. Δεύτερον, όπως σας υπέδειξα, θα ήθελα να μιλήσω για κάποιες παρεξηγήσεις που έχουν γίνει, ιδιαίτερα αυτές που σχετίζονται με το μοντέλο FASB. Άκουσα ότι κάποιοι προτιμούν το FASB εφόσον ε, δίνει από την πρώτη μέρα ζωής του τις αναμενόμενες απώλειες. Όμως είναι λάθος να αναφερόμαστε σε αυτές τις απώλειες ως απώλειες γιατί δεν είναι. Είναι απλώς ένα αριθμητικό αποτέλεσμα το οποίο κατασκευάζεται μέσω μιας ακατάλληλης, ε, ακατάλληλου συνδυασμού των εκτόσεων και των χρηματικών ροών. Δεν αναμένεται δηλαδή ε, τίποτα περισσότερο από την αναμενόμενη απώλεια που μπορεί να προκύψει στο ελληνικό χρέος εάν αφαιρέσουμε τις ε, τις αποδόσεις των ελληνικών ε, ομολόγων. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται όχι μέσω των τραπεζών, αλλά μέσω των κεφαλαικών αγορών. Επίσης, άκουσα ανησυχίες σε σχέση με το πρότυπο ε, IFRS, ότι εξαρτάται από υποκειμενικές εκτιμήσεις. Εξορισμό, όμως ένα μοντέλο για τις απώλειες, το οποίο θα υποστηρίζεται διεθνώς, θα πρέπει να συγκεντρώνει πληροφορίες από ένα μεγάλο αριθμό ε, ε, ε, στοιχείων. Επιπλέον, το IFRS 9 συμπεριλαμβάνει αυξημένες απαιτήσει αποκάλυψης των συγγείων, πράγμα το οποίο θα βοηθήσει τους επενδυτές να κατανοήσουν πώς ε, προετοιμάζονται, προετοιμάζεται η εφαρμογή των ε, προδιαγραφών, κάτι το οποίο δεν επιτρέπει τόσο ξεκάθαρο το, η προσέγγιση FASB. Τέλος, παραμένω να όσον αφορά την καταλληλότερα για την ε, λογιστική με δίκαιη ε, δίκαιο τρόπο και αξία. Καταρχήν από την αρχή, η, καταρχάς από την, εξ αρχής η ΕΚΤ είχε πει ότι δεν υπήρχαν τέτοιου είδους αποδείξεις, ότι δηλαδή ενδείξεις ότι το IFRS θα ήταν χειρότερο από το IS 39. Θα πρέπει να δούμε όμως πού ε, θα τεθεί η διαχωριστική γραμμή. Η εκτίμηση για το IFRS 9 σε σύγκριση με το IAS 39 ε, δίνει πιθανότητες και στις δύο προσεγγίσεις, ε, ενώ υπάρχουν και συγκεκριμένοι κίνδυνοι γιατί κάθε μια από τις δύο προσεγγίσεις, ε, καθώς το είδος των δραστηριοτήτων παίζει επίσης ρόλο, δανεισμός, εμπόριο, ε, holding ή πώληση. Επίσης υπάρχει από την έγκριση του IFRS 13 καλύτερη κατανόηση και χρήση των τεχνικών μέτρησης καθώς και διαφάνεια μεγαλύτερη, ιδιαίτερα όσον αφορά την υποκειμενικότητα των μετρήσεων. Σας ευχαριστώ και θα είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τους άλλους ομιλητές. Είναι οι απόψεις βέβαια όχι ομόφωνες θα τις χαρακτήριζα, αλλά κάποια ξεκάθαρα γενικά σημεία διαφάνηκαν Θέλω να ακούσουμε και συγκεκριμένα ε, τα συγκεκριμένα σχόλια για ένα συγκεκριμένο θέμα στο οποίο θα επανέλθω αργότερα. Θα ζητήσω από τον κύριο Βερό να κλείσει το μικρόφωνο του από την άλλη πλευρά. Πρώτος ομιλητής, πέντε λεπτά έχουμε για ερωτήσεις απαντήσεις. Τόλοχιαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας παρακαλέσω να ανταποκριθείτε στο αίτημα των κυρίων Γκίγκολτ και Καμάλ, δηλαδή να ζητήσετε τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Συγχρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για το IFRS 9, διότι έχουμε μια θετική ε, γνωμοδότηση από όλους τους σημαντικούς οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι Ευρωπαϊκές Αποπτικές Αρχές. Νομίζω λοιπόν ότι όπως προτείνουν οι συνάδελφοί μου είναι σημαντικό να έχουμε την νομοδότηση του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Τώρα, έρχομαι στο ερώτημά μου. Φυσικά το IFRS 9 είναι ένα θετικό βήμα σε σχέση με το 39. Γι' αυτό και είμαι και ευγνώμων στους εμπειρογνώμονες, τουλάχιστον τους περισσότερους που συμμερίζονται αυτήν την άποψη. Ωστόσο, υπάρχει ένα ζήτημα, αυτό που συζητείται περισσότερο και αφορά τη διαφορά μεταξύ του μοντέλ, των ΙΠΑ, σε σχέση με την καταχώρηση των απολειών, των ζημιών για το σύνολο του χρηματοπιστικού μέσου. Λογιστικό μοντέλο Η έκτα για το IFRS 9 προτείνει τρία στάδια. Πρώτο, για πρώτους, τους πρώτους 12 μήνες, αν επιδεινωθεί κατάσταση και στη δεύτερη φάση οι τράπεζες βέβαια τα ε, διάφορα που Το ερώτημά μου είναι, τελικά αυτή η διαφορά πόσο σημαντική είναι. Γιατί το FS 9 δίνει στις τράπεζες τη δυνατότητα να καταγράφουν ζημιές, απώλειες, αν βλέπουν ότι επιδεινώνεται τα μάλλη κατάσταση. Πόσο πια μεγάλη είναι αυτή η διαφορά, αυτό είναι το ερώτημά μου. Και απευθύνομαι σε όλους τους ειδικούς, ευχαριστώ. Ποιος θέλει να απαντήσει. Παρακαλώ, Άσλι. Καταρχάς, μια πρώτη απάντηση. Νομίζω προσπάθησα και να το πω. Υπάρχει μια διαφορά και αφορά τις διαφορετικές επιχειρηματικές πρακτικές ε, στην ε, Ευρώπη και στη ΣΥΠΑ και το ίδιο και τη λογιστική. Υπάρχει πολύ δανείο δοτική δραστηριότητα στη ΣΥΠΑ που δεν γίνεται μέσω του τραπεζικού συστήματος αλλά των κεφαλαίων αγορών που χρησιμοποιούν το μοντέλο fair value και νομίζω ότι υπάρχει ένα σοβαρό κίνδυνο και το είπα και πριν και δεν θα ήταν σωστό να μιλάμε για απώλειες ή ζημίες γιατί δεν πρόκειται για απόλυση. Και σε ένα ακαδημαϊκό σας σύγγραμμα νομίζω φέρεστε σε ό,τι αφορά αυτό το μέσο ως ένα ε, τεχνητό λογιστικό προϊόν αν το εφαρμόσετε σε ταμιακές ροές ε, και λάβετε υπόψη με όλα τα φαινόμενα αυτά, θα προκύψει απώλεια, θα προκύψει ζημία που δεν είναι όμως στην πράξη. Υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Ακόμη και με τις αναμενόμενες απώλειες για 12 μήνες, να υπάρξει πρόβλημα με τη δανειοδοτική δραστηριότητα γιατί μπορεί να μην μπορούν κάποιες επιχειρήσεις ε, να ε, προσαρμοστούν, γιατί θα πρέπει να καταχωρήσουν από την πρώτη μέρα τις απώλειες και να προσπαθούν μετά να τις αποσβέσουν. Έχει βρεθεί από τόσο συμβιβασμός. Επαναλαμβάνω όμω ότι μπορεί να επηρεάσει την οικονομική δραστηριότητα. Κάποιο μπορεί να πει ότι καλό θα ήταν ε, για να μην ε, φουσκώνουν τα βιβλία ε, τη τράπεζε. Αν δούμε το μοντέλο το αμερικανικό, εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει κίνδυνο περιστολή οικονομική δραστηριότητα και ιδίω αυτών που έχουν περισσότερο ρίσκο. Και δεν μιλάμε τι μεγάλε αλλά για μικρέ επιχειρήσει και αυτό με ανησυχεί. Επίση, τη ΣΥΠΑ είναι τελείω διαφορετική άποψη του κύκλου ζωή ε, lifetime. Αν δείτε και τη σχετική βιβλιογραφία, τρία με πέντε χρόνια είναι η προοπτική. Αυτό δεν είναι όμω ε, η πλήρη διάρκεια κύκλο ζωή. και αν δείτε τι έγινε ε, στι ΗΠΑ για τι ζημίε θα δείτε ότι υπάρχει ένας ανήρος συμβιβασμός ε, πριν από 15-20 χρόνια όπου η ΦΕΔ θέλησε και επέμεινε να έχει μεγαλύτερο αποθεματικό. Και το SEC το δέχτηκε. Αυτό λέω εγώ ανήρω συμβιβασμό. Ε, Ευχαριστώ, υπερμάς Μπερές. Αλλά μην ε, ξεπεράσετε τα δύο λεπτά στις ε, ερωτήσεις σας. Θα προσπαθήσω, κύριε Μπέρες. Τελευταία παρέμβαση μας δείχνει σε ποιο βαθμό τελικά για αυτά τα ζητήματα η προσέγγιση ε, των Ευρωπαίων μέσω αυτών των ε, προτύπων έναντι των είπα είναι ένα πρόβλημα και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Διάβασα πολύ προσεκτικά τις Μελέτε ή με απευθύνεται στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ε, δεν κατάλαβα ακριβώς τώρα που κολλάει αυτό, αλλά τέλος πάντων. Και δεν σημείωσα τίποτα ε, για την ε, απόρριψη του EFRS 9. Κάποια νοσταλγία την παρατηρώ βέβαια σε ό,τι αφορά τη λεγόμενη εύλογη αξία fair value, αλλά μάλλον θα πρέπει να λέγεται αγοραία αξία ε, και για την ίδια την ύπαρξη αυτών των προτύπων. Έχω κάποιες αμφιβολίες, αλλά εμείς θέλαμε το IFRS 9 για να λύσουμε ένα πρόβλημα που δεν θέλαμε να αντιμετωπίσουμε ουσιαστικά και το οποίο ήταν η εφαρμογή αυτής της εύλογης, η αγορά αξίας που θα έθετε σε κίνδυνο τα χρηματοδοτικά μοντέλα μας, ε, τα μοντέλα χρηματοδότησης της οικονομίας. Έχω δύο ερωτήσεις, γιατί κατάλαβα ότι υπάρχει μια πρόταση, μια σύσταση, δηλαδή να περιμένουμε να έχουμε από την ESB ε, τα πρότυπα και μετά να εξασφαλίσουμε μια ισότιμη μεταχείριση των δύο διαφορετικών προσεγγίσεων. Οι ασφάλειες ε, δεν βλέπω να θέλουν την ίδια ρύθμιση σε άλλους τομείς, αλλά τέλος πάντων ίσως να είναι κάτι συγκεκριμένο εδώ. Ποιος είναι ο κίνδυνος για τον τραπεζικό τομέα με την καθυστέρηση δηλαδή ε, της έγκρισης του IFRS 9 ε, σε σχέση με το τι κάνει το Συμβούλιο αυτό ε, για τη τεχνοτοπική σταθερότητα. Και το επόμενο μου ερώτημα είναι με βάση τους στόχους μας που είναι οι στόχοι για τη σταθεροποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών, ιδίω και με προοπτική την Ένωση Κεφαλαίων ποια είναι η θετική ή μη συνεισφορά του IFRS 9. Και βέβαια με τις ερωτήσεις μου κυρίως ε, απευθύνομαι στους υπέρμαχους και στους πολέμιους ε, των προτύπων IFRS 9, αλλά ο καθένας έχει την ελευθερία της άποψής του. Ο πρόεδρος βλέπω ότι ο κύριος Σεμπάρκο, κύριος και κύριος Βερόν, θα είναι το λόγο. Θα ήθελα να απαντήσω ε, στις ε, δύο ερωτήσει για το κατά πόσον το εργαλείο αυτό το άφηστερ 9 ε, θα πρέπει να ανασταλεί μέχρι να λυθεί το θέμα των ασφαλιών. Κοιτάξτε, κανείς δεν τάστη υπέρ αυτού, εγώ σίγουρα όχι και Όλοι οι άλλοι με τους οποίους έχω μιλήσει λένε όχι παρακαλούμε μην το αναστήλετε. Είναι ε, απαραίτητο το πρότυπο. Ήδη καθυστερήσαμε. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να ε, ορίσουμε μια ημερομηνία ταχύτατα που να ισχύει για τον τραπεζικό τομέα. Το θέμα είναι κατά πόσο αυτή η ημερομηνία θα ισχύει την ίδια στιγμή και για τον ασφαλιστικό τομέα, εκτό από τον τραπεζικό. Το ερώτημα που τίθεται είναι το εξή. Έχει νόημα να εφαρμόζει κανεί ένα κομμάτι του ισολογισμού τώρα και ένα άλλο κομμάτι μετά από δύο-τρία χρόνια. Αν έχουμε μία ολοκληρωμένη διαχείριση κεφαλαίων ή παγίων, ε, θα πρέπει και τα δύο πράγματα να τα κάνει κανεί την ίδια χρονική στιγμή. Γι' αυτό λοιπόν αυτή τη στιγμή υπάρχουν σκέψεις υπέρ του να επιτρέπεται μία επιλεκτική καθυστέρηση. Δηλαδή η αναβολή δεν θα είναι υποχρεωτική αλλά προαιρετική ε, και θα αφορά μόνο κάποιες ε, μονάδες, κάποια στοιχεία του ισολογισμού ενώ για όλα τα άλλα θα πρέπει να εφαρμόζεται το πρότυπο αυτό το συντομότερο δυνατόν. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο κύριος Μπάρκο σχετικά με την ταχύτατη εφαρμογή. Το θέμα των ασφαλιών είναι ε, πολύ εξειδικευμένο. Το εργαλείο FRS9 ισχύει για όλους τους τομείς. Άρα δηλαδή ε, οι ασφάλειες δεν μπορούν να κρατάνε όμοιρο αυτό το εργαλείο. Ε, θα πρέπει λοιπόν να συνεχιστεί η εξέλιξη χωρίς να παρεμποδίζεται αυτή η διαδικασία του χρηματοψηφιακού εργαλείου νέα. Κατά τα άλλα, όσον αφορά την αντιπαράθεση Ευρωπαϊκής Ένωσης με Ηνωμένες Πολιτείες, νομίζω ότι η μελέτη που κατατέθηκε στην ε, Επιτροπή Ακών είναι απόλυτα σαφής και συμφωνώ με το συμπέρασμα ότι η επιπτώση των διαφορών ανάμεσα στο IFRS 9 και των Αμερικανικών επιλογών δεν είναι σαφή αυτή τη στιγμή. Στην πρακτική εφαρμογή θα τα δούμε και δεν πρέπει να τα δούμε μέσα από το πρίσμα του συγκριτικού πλεονεκτήματος των Αμερικανικών τραπεζών έναντι των Ευρωπαϊκών τραπεζών. Εξακολουθούμε να μην γνωρίζουμε γιατί αποφάσισαν διαφορετικά οι Αμερικανικές τράπεζες, αλλά έχοντας ε, κατά νου το θέμα της σύγκλησης και του χάσματος νομίζω ότι θα ήταν πολύ περίεργο για την Ευρωπαϊκή Ένωση να αισθάνεται δεσμευμένοι από αυτά που γίνονται στις ε, Ηνωμένε Πολιτείε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εφαρμόσει το πρότυπο αυτό ε, στη δική της επικράτεια και να μην νιώθει κανένας είδους δέσμευση από αυτά που διαδραματίζονται στις Ηνωμένε Πολιτείε. Ο κύριος Καμάλ. Ευχαριστώ να ευχαριστήσω και όλους τους ομιλητέ μας. Έχω κανένα δυο γρήγορα θα προσπαθήσω ερωτήματα. Το πρώτο Γι' αυτό το μοντέλο αναμενόμενων ζημιών των 12 μηνών. Γιατί, γιατί 12 μήνες, ποια συλλογιστική υπάρχει πίσω από αυτό το 12 μήνο, γιατί τελικά ε, αν δούμε μετά από το μοντέλο, από το παράθυρο αυτό, ξέρουμε γιατί μιλάμε. Συμβιβασμοί, είπατε συμβιβασμοί, είναι κάτι που το ξέρουμε πολύ καλά και φυσικά δεν μπορούμε να πετύχουμε το ιδανικό μοντέλο. Έχετε εξετάσει μήπως άλλους συμβιβασμούς που θα οδηγούσαν ίσως όχι σε ένα μοντέλο της πρώτης ημέρας, ημέρας ένα, αλλά ένα άλλο μοντέλο. Όχι κατά ανάγκη της ημέρας ένα, της πρώτης μέρας. Να το δούμε αυτό ίσως ως επόμενο εφαλτήριο. Επόμενο ερώτημα είναι ουσιαστικά οι ανησυχίες μου για κάποια από τα σχόλια ε, ενός τέους μέρου του ISP, ο οποίο σε ένα ε, σύγγραμμά του που, έγινε σε ένα, που διαβάστηκε σε ένα συνέδριο της Ένωσης Λογιστών ε, και Ελεγκτών ε, και στην Ουαλία ε, αναφέρει κάποια πράγματα που διαγράφονται και τα οποία με εντυπωσιάζουν. Λέω ότι στον τομέα της χρηματοπιστωτικής πληροφόρησης ήταν απαραίτητο να είμαστε πιο διακριτική και οι Βρετανοί χρησιμοποίησαν πολλούς τρόπους να παρακάψουν την νομοθεσία που ε, χρειάστηκαν και το 2013 ώστε το παράνομα IFRS για τις ΜΜΕ να γίνει ένα νέο πρότυπο. Αυτά τα κάνουν, τα, αυτά τα λένε λοιπόν ακαδημαϊκοί. Και ο συγκεκριμένος έχει ε, επί δεκαετίες εργαστεί για τα πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Πώς μπορούμε εμείς ως βουλευτές να γνωρίζουμε τι οι ε, από την ΕΦΡΑΚ και από άλλους ε, υπεύθυνους για τη λογιστική που συνιστούν να υποστηρίξουμε το FRS 9 ότι έχουν δίκιο και ευσταθούν από νομικής πλευράς αυτά που υποστηρίζουν. Ευχαριστώ. Δεν είμαι νομικός, αλλά γιατί 12 μήνες ε, να απαντήσω αυτό το ερώτημα. Λέγεται σε αυτό το πρότυπο ότι από την αρχή καταγράφονται στη εύλογη αξία τα μετροπιστωτικά μέσα. Αυτό τι σημαίνει ότι εφαρμόζεται ε, το μοντέλο αναμενόμενων ζημιών ε, σε ο κύκλο ζωής Τώρα αυτές οι παρατηρήσεις που διαβάσατε έχουν να κάνουν μια διπλή καταγραφή γιατί βάζουμε 12 και όχι 24 και όχι 32 ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι ο λόγος τελικά ήταν ε, για να διατηρηθεί η ακαιρότητα μεταξύ ε, της δήλωσης ε, απόδοσης της τράπεζας για μια περίοδο, για ένα χρόνο και ταυτόχρονα να υπολογιστούν οι απώλειες ή μάλλον οι ζημίες ε, οι εκτιμόμενες για την ε, συγκεκριμένη αυτή περίοδο και να φαίνεται μια αναλογία ε, σε ό,τι αφορά το, την πιστοτική μερίδα και νομίζω ότι αυτή ήταν η επιλογή της προθεσμίας των 12 μηνών. Επίσης, δεν είναι το ίδιο με μια πραγματικά επισυμβήσα ε, ζημία. Αν εντοπίσουμε ότι υπάρχει ε, ε, αυτό το trigger, τότε φτάνεις και πιάνεις όλα αυτή τη χρονική περίοδο. Με βάση ένα συμβάν το οποίο έχει εντοπιστεί και το οποίο οδηγεί σε ζημίες. Κύριο Σάκερ. <clears throat> Κοιτάξτε, το επιχείρημα ότι σε τελική ανάλυση το, ο κίνδυνος, ο πιστοτικός καθορίζεται από το επιτόκιο, αυτό ισχύει για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ε, με την πάροδο των ετών, σε τελική ανάλυση, αλλάζει η φερεγγιότητα του υπόχρεου και ως εκ τούτου υπάρχει ένα αρχικό επιτόκιο το πραγματικό επιτόκιο το οποίο μπορεί κανείς ε, να διατηρήσει γνωρίζοντας ότι βεβαίως ε, αυτό το επιτόκιο συνοδεύεται και από κάποιους ε, κινδύνους. Τώρα, όσον αφορά αυτό το πρότυπο θα πρέπει ενδεχομένως να σκεφτούμε όχι τόσο το χρονικό διάστημα των 12 μηνών, αλλά πότε σε τελική ανάλυση θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι καταπίπτει η πίστοση. Όσον αφορά το αποτέλεσμα, νομίζω ότι ισχύει το ίδιο όπως και στο προηγούμενο χρηματοπιστωτικό εργαλείο, το 39. Έχουμε ένα δίκτυ για πιστωτικό γεγονός και από εκεί αρχίζει κανείς τους υπολογισμούς. Ε, αυτό ήταν στο 39. Τώρα, αυτό που είναι καινούριο στο IFRS 9 είναι ε, τα δύο πρώτα στάδια και εκεί λοιπόν θα πρέπει κανείς καταρχήν να δει τα προβλήματα. Το ένα είναι πως θα περάσουμε από το πρώτο στο δεύτερο στάδιο. Στην περίπτωση αυτή γίνεται μετάβαση αν επιδεινωθεί ουσιαστικά ο κίνδυνος ε, πιστοτικού γεγονότος. Αυτό μπορεί να ηχεί κάπως λογικό, αλλά στην περίπτωση αυτή δεν λαμβάνει κανείς υπόψη του πώς ξεκίνησε. Όταν υπάρξει ουσιαστική επιδείνωση μπορεί κανείς να πέσει από το πολύ καλό στο καλό. Τι γίνεται όμως αν από το ικανοποιητικό πέσει κανείς ε, στο επαρκές. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο θα πρέπει να σκεφτούμε κατά πόσον στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ε, διατηρήσουμε αυτό το σκεπτικό ή μήπως θα πρέπει να σκεφτούμε να λύσουμε το πρόβλημα έχοντας κατά νου το θέμα αρχής. Δηλαδή να ελέγχεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης κεφαλαίων. Άρα δηλαδή σε περίπτωση δανείου, ανεξάρτητα από τα αίτια ή οτιδήποτε άλλο, ε, να, ε, υπάρχει, να σκέπτεται κανείς το θέμα της φερεγκιότητας. Σε περίπτωση τέτοιας ε, επιχειρηματικές σκέψης, νομίζω ότι θα πρέπει κανείς περισσότερο να καταλήγει στο να μειώνει την αξία στους ισολογισμούς, τουλάχιστον αυτό έκαναν οι μικρές τράπεζες κατά το παρελθόν. Δηλαδή να σκεφτούμε κατά πόσο επιθυμούμε να διατηρήσουμε αυτή την επιχειρηματολογία ή μήπως είναι καλύτερα να βαδίσουμε με βάση το θέμα της αρχής. Δηλαδή η βελτίωση θα εγγράφεται στην περίπτωση όπου οι ίδιες επιχειρήσεις ε, τοποθετούνται για το θέμα της εξυπηρέτησης κεφαλαίων και στην περίπτωση αυτή ε, δεν είναι δυνατόν να εξοραίζονται ε, τα στοιχεία ε, απόσβεσης στους ισολογισμούς. Σε τελική ανάλυση, αν πρόκειται όμως για μεμονωμένα δάνεια, δεν μπορούμε από αυτά να εξάγουμε στατιστικά δεδομένα. Σε περίπτωση αμφιβολίας διαγράφεται η αξία εκείνη για την οποία δεν υπάρχει καμία εξασφάλιση. Και όλα αυτά πριν προκύψει πιστοτικό γεγονός με την έννοια του τρίτου σταδίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ξεκινήσω ευχαριστώντας τους ομιλητές που ήρθαν σήμερα και για τις ε, συμβολές τους στη συζήτηση μέχρι στιγμής. Τρει από εσάς είστε πολύ θετικοί, μιλάτε για τη σημασία για τις βελτιώσεις, λέτε ότι αξίζει να, να υιοθετηθεί, ότι είναι τεχνικός ε, ε συμπαγές το σύστημα κτλ. Όλα αυτά ακούγονται πολύ καλά και συμφωνώ μαζί σας. Όμως ο κύριος ε, Μπάρκ άρχισε να ρωτάει γιατί έπρεπε να κάνουμε αλλαγή. Γιατί αυτό ήταν η ανταπόκρισή μας ε, στην ε, πολύ έντονη κρίση ε, από το 2009. Αυτό είναι όλο. Χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο στα επόμενα χρόνια. Και η δεύτερη μου ερώτηση είναι πάντοτε υπάρχει θέμα ανάμεσα στο θέμα του κατά πόσο βασιζόμαστε στις αρχές ή στους κανόνες. Τώρα που βρισκόμαστε, γιατί συνήθως μετά από μια κρίση και οι πολιτικοί τείνουν να πηγαίνουν στους κανόνες, να βλέπουν αν αντιστοιχούν όλα σε αυτούς και μετά να θεωρούν ότι είμαστε ασφαλείς τέλος, για την ασφαλιστική, τον ασφαλιστικό τομέα ήδη έχουν τεθεί πολλά ερωτήματα σχετικά. Αλλά οι ασφαλιστικές εταιρείες που έχουν επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία δέχονται πολύ μεγάλες πιέσεις αυτή τη στιγμή. Δηλαδή την αντίθετη ερώτηση που, ρώτησε η συνάδελφος Μπερές. Είναι υπεύθυνο να τους επιτρέψουμε να έχουν μια μεταγενέστερη ημερομηνία ή μήπως θα έπρεπε να δραστηριοποιηθούν περισσότερο. Ποιος είναι ο κίνδυνος λοιπόν για ε, τον ασφαλιστικό τομέα. Σας ευχαριστώ. Νικολάς, ε, ζήτησες πριν το λόγο. Ναι, ήθελα να απαντήσω στην ερώτηση του κυρίου Καμάλα. εντάξει, μπορείτε. Θέλει κάποιος άλλος, κύριος Άσλεϊ, να πάρει το λόγο. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι αυτό αρκεί δεν νομίζω ότι υπάρχουν ενδείξεις, οποιασδήποτε ενδείξεις που να αποδεικνύουν ότι η λογιστική καταγραφή έπαιξε μεγάλο ρόλο στην προηγούμενη κρίση. Αλλά κατά πόσο μπορεί να βελτιωθεί και να βοηθήσει, ναι, εκεί ναι, το θεωρώ πως ναι, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ε, ζημιές ή τις αρνητικές επιπτώσεις. Πρέπει ωστόσο να προσέξουμε η Επιτροπή της Βασιλείας που κάνει καλή δουλειά για να επιτύχει την συνοχή να μην ε, καταλήξει στη θέσπιση τόσο πολλών κανόνων που τελικά να χάνει την ουσία της η αρχή ε, την οποία επιθυμούμε να εφαρμόσουμε. Τώρα για τις ασφαλιστικές εταιρείες ε, πιστεύω πάλι πως είναι θετικό αυτό το πρότυπο, αλλά δεν θα λυθεί το θέμα, το πρόβλημα της ασφαλιστικής βιομηχανίας και η διαφάνεια που μπορεί να απέλθει μέσω του FRS 9 σε αυτόν τον τομέα ε, σημαίνει ότι θα πρέπει να εκπονηθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα και το πρότυπο για τις ασφαλιστικές. Εάν δεν κάνουμε κάτι δηλαδή ε, για το παθητικό κομμάτι του ισολογισμού, ε, τότε δεν θα ε, δούμε τον αντίκτυπο των εντάσεων και των πιέσεων που δέχεται τώρα ο ασφαλιστικός κλάδος. Ευχαριστώ. Ο Φάμπιο Ντεμάζη. Θα ήθελα να διαφωνήσω με την προελίσσα ότι εδώ δεν υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις. Κάθε άλλο, έχουμε διαπιστώσει ότι σε πάρα πολλά πιστοτικά συστήματα όπου η χορήγηση δανείων εξαρτάται όλο και περισσότερο από εξασφαλίσεις, ε, όταν υπάρχει υπερβολική ζήτηση διαπιστώνουμε υπερθέμανση και στην αντίθετη περίπτωση ε, διαπιστώνουμε μια αρνητική εξέλιξη. Άρα δηλαδή είναι σημαντικό το ότι το επιτόκιο προσαρμόζεται στον πιστοτικό κίνδυνο αλλά το επιτόκιο δεν είναι κάτι το εξωγενές. Ε, το επιτόκιο ε, σε περίπτωση αμφιβολίας οδηγεί ε, ή εξαρτάται από την φερεγγιότητα του υπόχρεου. Όταν ε, ο υπόχρεος δεν είναι φερέγγιος, ε, αυξάνεται το επιτόκιο. Τέλος πάντων, θα κάνω κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις προς τον κύριο Χάκερ. Συγκεκριμένα, θεωρείται ο κίνδυνος ε, η διακριτικότητα που υπάρχει στο IFRS 9 σχετικά με, τα προβλεπόμενα, με τις προβλεπόμενες ζημιές αυτή η εχεμήθεια θα οδηγήσει στο ότι να υπάρχει καθυστέρηση από την πρώτη φάση τη δεύτερη φάση η οποία θα γίνεται και επιλεκτικά. Πιστεύετε ότι υπάρχει κίνδυνος ακριβώς αυτή η αχεμήθεια να οδηγήσει στα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίσαμε στο IFRS 39 και στην περίπτωση αυτή η αναγνώριση των ζημίων θα οδηγήσει σε σημείο από το οποίο δεν μπορεί κανείς πλέον να επανέλθει, άρα δηλαδή θα φτάσουμε σε ύφεση. Απάντηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς, η απάντησή μου θα είναι κάπως γενική. Τίθεται το ερώτημα κατά πόσον το χρηματοψηφιστικό αυτό πρότυπο αποτελεί βελτίωση ή όχι. Νομίζω, συμφωνούμε όλοι, ότι όσον αφορά την εγγραφή στο ισολογισμό του fair value, value ε, της θεμητής αυτής αξίας, δεν έχουν αλλάξει και πάρα πολλά. Περίπου κάπως έτσι ε, είναι τα πράγματα και αν το πρόβλημα ήταν το fair value, ε, το IFRS e 9 στην περίπτωση αυτή ε, έχει την ίδια αποτελεσματικότητα όπως το 39, άρα δηλαδή και εγώ δεν ρωτώ με ποια είναι η αποτελεσματικότητά του. Η μόνη ουσιαστική διαφορά είναι αυτό το μοντέλο μείωσης της αξίας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έχουμε και πάλι μία ε, αιτιολογική προσέγγιση. Βεβαίως η αναζήτηση των αιτίων ε, είναι πάντα συμπαθική γιατί στην περίπτωση αυτή ε, υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι κανόνες αλλά υπάρχει και ένα μεγάλο περιθώριο εκτιμήσεων έννοιες ε, όπως ε, ουσιαστική επιδείνωση εκεί υπάρχει μεγάλο περιθώριο ελιγμών. Μπορεί κανείς να ε, ζητήσει καθυστέρηση, αλλά σε τελική ανάλυση ισχύει το εξής. Σε περίπτωση μείωση της αξίας πάντα υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας και λήψη αποφάσεων κατά το δοκούν. Μόνο που κατά την άποψή μου χρειαζόμαστε προσανατολισμό με βάση την αρχή το τι ισχύει, γιατί αυτή η αναζήτηση των αιτίων δεν λύνει το πρόβλημα. Οποτεδήποτε υπάρχουν κανόνες, όπως παραδείγματο χάρη ουσιαστική επιδείνωση, προηγουμένω, υπενήχθην ότι αυτό καθαρά λογικά δεν είναι σημαντικό. Αυτό που έχει σημασία είναι στη τελική ανάλυση ποια είναι η κατάσταση του υπόχρεου στο τέλος και όχι εκ των προτέρων στην αρχή αυτό που σημαίνει στο τέλος. Αυτό είναι το καθοριστικό. Άρα δηλαδή το κριτήριο που χρησιμοποιείται είναι τροτό... Ε, περιέχει κάποιο περιθώριο διακριτικής ευχέρειας και το μόνο που μπορεί να βοηθήσει είναι να προχωρήσουμε με μία προσέγγιση λειτουργώ με βάση την αρχή. Αυτή την προσέγγιση. Η, τα λογιστικά πρότυπα άμεσα ή έμεσα επηρεάζουν την ε, συμπεριφορά επί του κινδύνου και στη τελική ανάλυση ισχύει το εξής. Αν μπορεί κανείς να παρακάμψει κάποια κριτήρια, όπως ας πούμε το θέμα του σημαντική επιδείνωση ή όχι, ε, υπάρχει πάντα το κίνητρο της καθυστέρησης. Το πρόβλημα είναι όχι το τι θα κάνουμε σε περίπτωση κρίσης, αλλά το κατά πόσον η ίδια η λογιστική, τα λογιστικά πρότυπα με οδηγήσουν στην κρίση. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει εκ των προτέρων να έχουμε προβλέψει κάποιες ζημιές ε, με συγκεκριμένα μοντέλα, ας πούμε με το fair value, έχουμε κάποιες δυνατότητες να μετακινηθούμε προς τα πάνω. Αν έρθει όμως η κρίση υπάρχει η παγίδα που είναι πολύ πιο έντονη και εκεί υπάρχει το κίνητρο ακόμα πιο έντονο, το κίνητρο της μετάθεσης. Ναι, πράγματι υπάρχει διακριτική ευχέρεια. Ε, σε περίπτωση κρίσης το IFRS 9 ε, είναι καλύτερο από το 39, αλλά επαναλαμβάνω σε περίπτωση κρίσης εξακολουθεί να είναι αρνητικό, να είναι κακό. Καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω για την ακρόαση αυτή που διοργανώσαμε γιατί είναι σημαντικό το θέμα. Να κάνω καταρχάς μια μεθοδολογική παρατήρηση. Ένα μεγάλο πρόβλημα για εμάς ως νομοθέτες, νομίζω τουλάχιστον, είναι ότι νομοθετούμε για την ουσία Πολύ δύσκολα όμως μπορούμε να έχουμε μια ε, γνώμη επίσημη, ειδική, από κάποιον που δεν έχει όμως σύγκρουση συμφερόντων. Ένας για 15 ήταν ε, ηγέτες του Κέντρου Αριστείας με την Deloitte για τα πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, ένας με την KPMG για πολλά χρόνια και τώρα είναι στο ε, Διοικητικό Συμβούλιο της ε, γνωστής Barclays Bank. Όχι ότι είναι προσωπικό το ζήτημα, δεν το κρίνω εγώ και ότι και θέλω. Απλά λέω, δημιουργείται ζήτημα. Έχουμε δύο άτομα εδώ που έχουν στενή σχέση με την ΕΦΡΑΚ και ταυτόχρονα έχουν αυτό το επαγγελματικό παρελθόν. Και πολύ λίγες φωνές στον ίδιο αυτό οργανισμό είναι ανεξάρτητες. Και αυτό εμένα μου δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα. Ερώτηση τώρα προς τον κύριο Μπάρκο. Η G20. Ο κύριος Το 2009 δημοσίευσα μια έκθεση. Ορίζοντας κάποια κριτήρια για το τι πρέπει να γίνει με τα νέα λογιστικά πρότυπα. Δεν θέλω να τα καταγράψω και να τα αναφέρω όλα. Αλλά το πρώτο λέει να περιοριστεί η πολυπλοκότητα των λογιστικών ε, προτύπων για τα χρηματοπιστωτικά μέσα. Και τώρα πρέπει να τα πω γερμανικά. Τι γράψα το 14, κύριε Μπάρκο. Από την αρχή ήταν ο στόχος να μειωθεί η περιπλοκότητα και σήμερα βεβαίως κανείς πια δεν μιλάει γι' αυτό. Θα μπορούσατε κύριε Μπάρκο να σχολιάσετε. Η G20 τελικά ή μάλλον το IFRS 9 αν κατάφερε να πετύχει ε, αυτό που ζητούσαν οι G20 και για τον κύριο Χάκη που κάνετε συγκεκριμένε προτάσεις και λέτε μπορείτε να το εγκρίνετε αλλά να έχετε κάποια caveat. Τι θέλετε να ε, και γιατί τι πρέπει να αποφύγουμε. Thank you, Please. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να σχολιάσω παλιότερα αυτά. Τέλος πάντων, ε, αυτό που, ζήτησαν, ε, που ζήτησε η ομάδα των 20, το G20, για το ε, περιορισμό τη πολυπλοκότητας στα χρηματοπιστωτικά μέσα είναι σωστό αίτημα, αλλά δεν ήταν και ποτέ στόχος, αυτός σκοπός αυτός. Πάντα πρέπει να το συσχετίσουμε με όλους τους άλλους παράγοντες. Όταν ξεκίνησε τη διαδικασία το 2008 και την προηγούμενη χρονιά, ε, από το αίτημα αυτό δηλαδή. Θέλαμε, ε, είχαμε ένα γενικό σχέδιο 20 σελίδων που όμως έγινε πολύ πιο ογκώδε σιγά σιγά λόγω των ζητημάτων που έπρεπε να αντιμετωπιστούν και γιατί τώρα έχουμε ένα νέο μοντέλο απομείωσης αξίας που φαίνονταν να το γνωρίζουν από τις οπτικούς κανόνες ήδη, αλλά έπρεπε να το εξηγήσουν και αυξήθηκε ακόμη περισσότερη βιβλιογραφία και για αυτό το λόγο. Άρα η πολυπλοκότητα, ναι μεν δεν έχει αντιμετωπιστεί επαρκώς, αλλά ε, δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι μπορεί να αντιμετωπιστεί ποτέ επαρκώς. Δεν μπορώ να φανταστώ ένα πρότυπο που έχει να κάνει με χρηματοπιστωτικά μέσα και να μην είναι ε, λιγότερο από 20 Ο David Tweety θα μπορούσε να τα πει ανάποδα. Διάβασε το iStudy 9 αν, ήταν δεν θα, αν δεν ήταν ειδικό δεν θα καταλάβαινε. Ή αντίστροφα, αν κάποιο μπορεί να γράψει ένα πρότυπο για τα χρηματοψηφιακά μέσα και να μην υπερβεί τι 20 σελίδε, μάλλον δεν έχει καταλάβει γιατί μιλάμε. Μα είναι 20 σελίδε πιο μακροσκελέ. Όχι απλά 20 σελίδε, έγινε ακόμα πιο πολύπλοκο. Άρα άλλε 20 σελίδε παραπάνω. Αυτό λέω, λέει ο κ. Κίκολτ. Ναι, συμφωνώ, αλλά δεν θα κολούσα τόσο πολύ στις 20 επιπλέον αυτές σελίδες. Νομίζω ότι μπορείτε να συμφωνήσετε ότι 500 σελίδες να είναι ένα πολύ μακροσκελές. Τώρα 500 ή 520 δεν είναι πια και τόσο τεράστια διαφορά. Αλλά συμφωνούμε νομίζω ότι να είναι μακροσκελές. Ο Νίκολας είχε ζητήσει το λόγο. Γρήγορα παρακαλώ. 30 δευτερόλεπτα μήπως. Ακούστε δύο πράγματα. Ή μάλλον ένα σε ό,τι αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων ήταν ένα θέμα το οποίο έθεσε ο κύριο Καμάλ και ο κύριο Γκίγκολ πολύ σωστά. Είναι εύκολο βέβαια εγώ να τα σχολιάζω γιατί ποτέ δεν ήμουν εξαρτημένος είτε από τους ε, τέσσερις μεγάλους ε, αλλά ε, πρέπει να ξέρετε, υπόψη σας ότι το Ινστιτούτο μας έχει ασφαλιστικές δικλείδες και χαίρομαι που μπορώ να συμμετέχω σε αυτή τη συζήτηση, γιατί δεν νομίζω ότι μόνο η κλειστή λογιστική κοινότητα θα πρέπει να συμμετέχει. Ξέρω ότι υπάρχουν διαφορετικέ διαφορετικές σε αυτό το κύκλο των λογιστών και στην ΕΦΡΑΚ. Ε, γενικά υπάρχει μια τεταμένη συζήτηση, έντονη συζήτηση. Ε, σίγουρα και από οικονομικέ πλευρέ και από άλλες πλευρές ε, το ΕΦΕΣ. Το ε, επηρεάζουν οι Big Four, οι μεγάλοι τέσσερις. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Αλλά σίγουρα είναι σημαντικό να ακούσετε από διάφορα επιχειρήματα για το IFRS 9 και να μπορέσετε να καταλήξετε σε μια περιστατωμένη άποψη. Η Μπάρμπαρα Κάπελ, ο πρόεδρος δεν είναι στην αίθουσα, δεν τη βλέπω. Ο κύριος Σόλο για να έχει το λόγο. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το ερώτημά μου τώρα ή μάλλον σχόλιο, όπως θέλετε, πάρτε το. Με εξέπληξε κάπως, ανέ, ναι, συγγνώμη που απομακρυνθήκα από το μικρόφωνο, ε, με απογοήτευσε κάπως το γεγονό ότι το ICB e για το IFRS 9 έχει δαπανίσει πολύ χρόνο. Εργάζεται εδώ και καιρό για αυτό το πρότυπο. Και, το ΕΦΡΑΚ όμως δεν μπορεί να επηρεάσουν ε, σε ό,τι αφορά δηλαδή, την μελέτη αντικτύπου, ε, πολύ λίγα μπορούν να πούν. Προσπαθώ να βρω για αυτό το πρότυπο, προσπαθώ να βρω κάποια αριθμητικά στοιχεία. Αλλά οι εκτιμήσεις δεν ξέρω πού βασίζονται. Σας ρωτώ λοιπόν, εσείς τι πιστεύετε. Ε, η ΕΚΤ και η ΕΦΡΑΓ θα πρέπει να επενδύσουν μέσα και πόρους για αυτή τη μελέτη αντικτύπου. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε συνηθίσει τις μελέτες αντικτύπου για τους κανονισμούς που εγκρίνουμε εδώ. Ευχαριστώ. Thank you. Uh, Mr. Yes, Mr. Ashley. Can I try and respond to that, that last point and, and possibly not totally uh, convincingly, but Λοιπόν, κοιτάξτε, θέλω να πω το εξή ότι οποιαδήποτε αξιολόγηση επιπτώσεων ή αντικτύπου θα πρέπει σε κάποιο βαθμό να είναι ποσοτική για να μπορεί κανείς να κατανοήσει ποιες είναι οι επιπτώσεις. Παραδείγματο χάρη όσον αφορά τη ζημιά, το impairment, ε, τι ύψου είναι. Ε, πρέπει να το ξέρει κανείς ε, για να γνωρίζουν και οι άνθρωποι τι να απαντήσουν. Το πρόβλημα τόσο για τον ISB και για τον ΕΦΡΑΚ είναι ότι προσπάθησαν να πείσουν την, τις τράπεζες να παρουσιάσουν αναλύσεις αλλά δεν έγινε αυτό. Και δεν έγινε γιατί δεν είναι εύκολο να εφαρμοστούν τα πρότυπα. Δεν είναι κάτι που στρέφεται κανείς αυτό και αρχίζει να παράγει αριθμούς. Ας πούμε η δική μου η τράπεζα, η Barclays, εμείς έχουμε ένα project ε, που περιλαμβάνει 250 ανθρώπους για 2,5 χρόνια για να εφαρμόσουν το IFSR 9. Μιλάμε για τέτοιου είδους κλίμακες. Είναι λοιπόν πολύ δύσκολο κάτω από αυτές τις συνθήκες να κάνει κανείς κάτι άλλο πέρα από το να προσφέρει ε, σενάρια υψηλού επίπεδου όσον αφορά τις επιπτώσεις. Αυτή είναι η πραγματική δυσκολία. Δεν ξέρω αν σας βοηθάω στο να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα, αλλά εν πάση περιπτώσει ε, είναι και κάτι που δεν λύνεται και πολύ εύκολα. Άλλος παρακαλώ, μήπως επιθυμεί κάποιος άλλος ε, να πει κάτι. Ο κύριος Χάκα. Κοιτάξτε, ε, υπάρχει ακόμα το ερώτημα του κυρίου Γκίγκολτ που νομίζω ότι δεν έχει απαντηθεί, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένα πράγματα που ελέγχθησαν. Λοιπόν, Υπάρχει εδώ μια σύγχυση. Πολλοί λένε ότι ζούμε σε ένα περίπλοκο κόσμο. Ε, Βεβαίω και τα χρηματοπιστωτικά είναι πολύ μπερδεμένα. Αλλά σε τελική ανάλυση δεν πρέπει κανείς ε, να τα ε, συγχαίει με τα μη επιλύσιμα. Είναι δύσκολα, αλλά δεν είναι μη επιλύσιμα. Εγώ τώρα δεν θέλω να κάνω διαφήμιση των δικών μας των προτύπων, αλλά εν πάση περιπτώσει σε λίγες μονοσελίδες και σε λίγα, λίγες παραγράφους μπορεί κανείς να αναζητήσει τη λύση. Υπάρχει βέβαια σχολιασμός, αλλά σχολιασμός σε τελική ανάλυση σημαίνει ε, ποικιλία απόψεων. Έγινε λόγος για τη σύγκρουση συμφερόντων ε, και πρέπει ε, να έχει κανείς κατά νου την ιστορία αυτού του οργανισμού ε, που ασχολείται με τα λογιστικά πρότυπα και αν δει κανεί λιγάκι και το βιογραφικό των ανθρώπων που υπάρχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτού του Οργανισμού Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, αν δει κανεί αυτά τα βιογραφικά δεν θα εκπλαγεί για το ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν σκέφτονται με βάση την αρχή. Όσον αφορά αυτό που ρώτησε ο κύριο Γκίγκολτ, το 2009 είχε δοθεί η υπόσχεση επεξεργασίας και εγώ είχα προβλέψει τότε ότι θα επεκταθεί το περίφημο fair value. Εγώ επιμένω σε αυτά που έχω γράψει και κατά το παρελθόν. Ο κύριος Γκίγκολτ ρώτησε τι πρέπει να γίνει. Έχω λοιπόν το εξής πρόβλημα. Αν τώρα πω μην εγκρίνετε το πρότυπο, κατανοώ ότι δεν ξέρω το πρότυπο αυτό ε, ψήνεται, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, εδώ και πέντε χρόνια. Εμπειρογνώμονες ε, τελικά ε, το έχουν αποδεχτεί, ε, τα μηχανογραφικά έχουν προσαρμοστεί σε αυτό το πρότυπο. Αν δεν εγκριθεί λοιπόν θα έχουμε να κάνουμε με μια καταστροφή. αν θέλετε θα έχουμε να κάνουμε με μια κατάσταση που επικρατεί στην κατασκευή του αεροδρομίου του Βερολίνου το γεφύρι της Άρτας εν ολίγη στα ελληνικά. Όσον αφορά λοιπόν το fair value, ε, κατ' ουσίαν έχουμε να κάνουμε ακριβώς με το ίδιο πρόβλημα. Δηλαδή, αν θεωρεί κανείς ότι είναι σοβαρός οργανισμός, βεβαίως και υπάρχουν ε, δημοκρατικές διαδικασίες, ε, άρα δηλαδή κάτι πρέπει να γίνει και υπάρχουν ορισμένοι τομείς όπου δεν θα δημιουργείται πρόβλημα αν δεν ενεκρίνεται αυτό το εργαλείο. Στη τελική ανάλυση, αυτό το fair value ε, με βάση το πρότυπο 9 θα πρέπει να εντάσσεται στους ε, ισολογισμούς ε, σε περίπτωση όπου οι πληρωμές έχουν οριστεί στα συμβόλαια. Αλλιώς ε, οτιδήποτε ξεφεύγει από αυτό ε, μπαίνει ε, στον ισολογισμό ζημιών και κερδών. Βεβαίως θα πρέπει κανείς να διερωτηθεί μία εταιρεία περιορισμένης ευθύνης γιατί να πρέπει και αυτή να χρησιμοποιεί αυτήν την fair value. Στην μείωση της αξίας, το είπα και προηγουμένως, έτσι θα το πω και τώρα πολύ πρόχειρα, θα πρέπει να ισχύει ένας κανονισμός ε, που θα υπερισχύει των αιτιολογικών αναζητήσεων. Δηλαδή να μην ζητάμε από τις επιχειρήσεις ε, σε τελική ανάλυση να εφαρμόζουν στα λογιστικά πρότυπα ε, θέματα αρχής και μετά να γίνεται απόκληση από αυτά. Σας είπα ότι σε μεμονωμένα δάνεια δεν υπάρχει κάποια δυνατότητα να υπολογίσουμε στατιστικά κάποια στοιχεία. Άρα δηλαδή αυτές είναι δύο αλλαγές. Η μία είναι ότι ε, βασιζόμαστε σε επίπεδο αρχής ε, στην μείωση της αξίας και το δεύτερο είναι ότι σε ορισμένους τομείς ξεκινάμε από το fair value, κάτι που δεν θα δημιουργήσει κανένα πρόβλημα στην εγγραφή στο, στους ισολογισμούς. Η κυρία Περβάνς Περές. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω αυτή τη φορά τον κύριο Χάκερ. Γιατί πολλές από τις επικρίσεις που εσείς διατυπώσατε είναι επικρίσεις που γνωρίζω από το που ασχολούμαι με αυτά τα θέματα, δηλαδή εδώ και αρκετό καιρό. Αλλά το ζήτημα δεν είναι να ξέρουμε πώς λειτουργεί το, ε, το, το IASB, ποια είναι τα προβλήματα κτλ. Το θέμα είναι τι κάνουμε με την απάντηση που μας έδωσε το IASB στην ερώτηση όπου επικρίνουμε το fair value και εσείς μας λέτε μείναμε στην ίδια κατάσταση. Η ερώτησή μου είναι λοιπόν, προτιμάτε να μείνουμε στο, 39, στο IRS 39 ή να μπούμε στο IFRS 9, αν είχαμε να διαλέξουμε αυτά τα δυο. Εσείς προτιμάτε το ε, IAS 39. Και μια ερώτηση για τον Νικολά Βερό. Πώς μπορούμε να πούμε ότι μένουμε στην υπόθεση Μπαϊού, στο ΙΕΦΡΕΣ 9, όταν είναι πιο περίπλοκο σε τρεις κατηγορίες, ειδικά για να ξεφύγουμε σε μεγάλο βαθμό από αυτή τη λογική της, ε, αγορά, της αξίας της αγοράς, όπου θεωρούμε ότι δεν χρειάζεται να υποβάλουμε όλα μας τα τραπεζικά συστήματα. Ευχαριστώ. Κύριε Χάκερ πρώτα. Όχι πολύ ώρα παρακαλώ γιατί Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε, η κριτική αυτή για το fair value είναι πολύ πιο παλιά. Από το 1848 απαγορεύτηκε αυτή η αξιολόγηση. Βλέπετε επαναλαμβάνεται η ιστορία. Όσον αφορά το fair value, το τι πρέπει να γίνει. Κοιτάξτε, αν θέλω να κάνω πραγματικά ριζοσπαστικές προτάσεις, τα έλεγα ότι εγώ ε, δεν συμφωνώ με αυτό το θέμα των προτύπων, αυτό όμως είναι μακροπρόθεσμο. Το θέμα είναι τι μπορεί να γίνει βράχη πρόθεσμα. Αν δεν υιοθετήσουμε το IFRS 9, τότε θα εξακολουθεί να ισχύει το IFRS 39 ε, ή αν θέλετε ε, κάποια στοιχεία του FRS 9 που έτσι κι αλλιώς εφαρμόζονται στην αγορά. Αν θέλετε να αλλάξετε κάτι, ε, τότε αυτή τη στιγμή είναι η κατάλληλη στιγμή για να εξαιρεθούν κάποιες ρυθμίσεις ε, και μακροπρόθεσμα. Θα πρέπει κανείς να πει στο ISB ότι θέλουμε μία στάνταρτ ε, κάποιους στάνταρς ε, υπολογισμούς και στάνταρ πρότυπα ε, ίσως ε, θα μπορούσε κανείς να τα αναθέσει αυτά σε κάποιους ιδιώτες. Αλλά σας λέω και πάλι, αυτά γίνονται μόνο μακροπρόθεσμα. Βράχει πρόθεσμα, θα πρέπει κανείς να δει με μονομένους κανονισμούς, να εντοπίσει πού ακριβώς βρίσκονται τα προβλήματα, τι έχει λυθεί και να σκεφτούμε κατά πόσον θα πρέπει όλα αυτά να γίνουν αποδεκτά ή όχι. Πολύ ωραία, αλλά ξέρετε το ερώτημα ήταν συγκεκριμένο τι θέλετε, το 39 ή το 9, ποιο από τα δύο προτιμάτε. Αυτή ήταν η ερώτηση με απλά λόγια. Εντάξει, εσείς τα σώτασεστε υπέρ ενό διαφορετικού μοντελού, ούτε 9 ούτε 39, αλλά κυρία Πέρας λέει τι θέλετε, το 9 ή το 39. Συγγνώμη, αλλά δεν κατάλαβα πολύ καλά το ερώτημα. Μήπως η κυρία Μπερές θα μπορούσε να τα επαναλάβει. No, but, Mr. Um, Hacker said... Ο κύριος Χάκερ λέει ότι με το IFRS 9 ε, παραμένουμε στην εύλογη αξία. Το fair value συμφωνείτε. Δεν έχει εξαφανιστεί το fair value από το IFRS από το πλαίσιο αυτά για τα χρηματοπιστωτικά μέσα. Άρα, επ' αυτήν την έννοια πράγματι δεν απαλήφεται. Μπορούσε να πει κανεί ότι έχουμε κολλήσει ε, σε αυτό. Αλλά αυτό δεν το θεωρώ κακό, αλλά καλό χαρακτηριστικό του συστήματος γιατί ε, χρειαζόμαστε ε, τα market values. Αλλιώς θα υπάρξει μεγάλο ποσοστό χειραγώγησης από τις αγορές. Πάνω από 8 χρόνια κράτησε η χρηματοπιστωτική κρίση στην Ευρώπη και πολύ περισσότερο πληγήκαμε από την χειραγώγηση ε, από τους τραπεζίτες που προσπαθούσαν να καλύψουν τις ζημιές τους παρά από προκυκλικές επιπτώσεις ε, σε σχέση με το fair value. Άρα νομίζω τώρα έχουμε πιο μεγάλη εμπειρία από ό,τι είχαμε όταν πρωτοξεκινήσαμε το 2008 ή 2009 την όλη συζήτηση και το πρόβλημα με την κρίση δεν ήταν η ευλογιαξία αξία το fair value αλλά η ανεπαρκής λογιστική καταγραφή από τους τραπεζίτες που θέλανε να κρύψουν τις απώλειε, τι ζημιές τους. Ό,τι αφορά το πρώτο ερώτημα της κυρίας Μπερέσα. Ε, για τα carve-outs θα ήθελα να κάνω ε, ένα σχόλιο. Δεν επιτρέπεται το carve-in από τον κανονισμό. Δεν ξέρω κατά πόσο επιτρέπεται και το carve-out. Αυτό είναι ένα νομικό ερώτημα. Δεν έχει βέβαια υπάρξει απόφαση δικαστηρίου, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι ε, μπορούμε να κάνουμε αυτό το carve out. Ε, δεν θεωρώ ότι ευσταθεί πολύ όμως ε, ως ε, ισχυσμός. Επάνω στο fair value τώρα. Νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο στο πλαίσιο της αξιολόγησης του κανονισμού IAS που έκανε η Κομισιόν πέρυσι. Εκεί η Επιτροπή μελέτησε τη βιβλιογραφία ε, για το πώς επηρέασαν τα λογιστικά πρότυπα ε, την κρίση. Και πρέπει οι βουλευτές νομίζω να διαβάσουν αυτό το έγγραφο που περιλαμβάνεται ως παράρτημα στην έκθεση αξιολόγησης. Είναι ποιοτικό έγγραφο. Και σε αυτή την αθρότητα της βιβλιογραφίας αναφέρεται ακριβώς οτιδήποτε έχει υποθεί από τον οποιονδήποτε, οπουδήποτε για αυτό το ζήτημα. Και πραγματικά είναι στριπτικά τα στοιχεία. Δηλαδή δεν φταίει η λογιστική του Fair για το τι έχει υποφέρει τα τελευταία χρόνια και πάμε και πιο πέρα ο τραπεζικός τομέας. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Θα σας δώσω το λόγο, κύριε Χάκερ. Αλλά και εγώ έχω μια ερώτηση. Από τι κατάλαβα, πρώτον, συμφωνούν όλοι ότι έχουμε ένα πρόβλημα με τις ασφάλειες. Γιατί δεν συμπίπτει η έναρξη ισχύω του νέου FRS 4 και άρα έχουμε αναντιστοιχεία στο λογιστική ενεργετικού παθητικού. Όλοι νομίζω συμφωνούμε ότι αυτό το πρόβλημα πρέπει να λυθεί. Οπότε καταλαβαίνω με δύο τρόπους μπορεί να λυθεί. Και ο πρώτος μου φαίνεται πιο λογικός δηλαδή για τις ασφάλειες να έχουμε μια καθυστέρηση της έναρξης ισχύω μέχρι ότου ε, και το άλλο σκέλος τεθεί σε ισχύ. Υπάρχει όμως και μια άλλη λύση να εφαρμόσετε ο, ο σαν να. Δεν ξέρω αν αυτό ε, σας βρίσκει συμφωνούσε. τι μπορούμε να κάνουμε με κάποιες υποεπιλογές για τη βασική επιλογή. Όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να επιληφθεί το πρόβλημα. Και δεύτερον, Από ό,τι κατάλαβα αληθεύει ότι δεν είναι το μονέτιο της κρίσης στον τραπεζικό τομέα, το fair value. Όμως ίσως υπάρχει κάποια προκυκλικότητα. Με το fair value δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να αμφισβητηθεί εύκολα. Αυτό τώρα ε, γίνεται, με αυτό το πρότυπο γίνεται ένα βήμα προς τα εμπρός και όχι προς τα πίσω. Γιατί κάτι τέτοιο δεν θα ήταν καλό και δεν συμμερίζονται και την άποψη του Νίκ. Τι πρέπει να γίνει με το φερβάλιο, Νίκ λέει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεν ε, χρειάζεται να το απαλείψουμε. Το θέμα είναι τι κάνουμε από εδώ και πέρα για να αντιμετωπίσουμε τις ελλείψεις και τις αδυναμίες που είδαμε. Δεν προσπαθώ να λήξω σε συμβιβασμό των διαφορετικών σας απόψεων, γιατί βλέπω ότι διαφωνείτε. Απλά πώς τη βλέπετε αυτή την προσέγγιση, έχει κάποια λογική. Ποιος θέλει να ξεκινήσει. Hacker. Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ ε, ξέφρασα την κριτική μου και αμφισβητώ θέλω να σας πω ότι θα αυξήσει την διαφάνεια το fair value και ότι οι ζημιές που θα προκύψουν ε, στην εγγραφή στους ισολογισμούς ότι αυτές μπορούν να αποφευχθούν με το fair value. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτά. Με πάση περιπτώσει, μπορείτε να σκεφτείτε το τι θα κάνετε. Όπως ε, σας είπα, ε, ανέφερα δύο σημεία όπου μπορούν να υπάρξουν κάποιες αλλαγές και ξέρετε κάτι, τώρα σε αυτή τη φάση δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Αυτά. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να φερθώ στο πρώτο σας ε, ερώτημα αν θα υπάρξει καθυστέρηση ή όχι, αναβολή ή όχι. Νομίζω ότι ετέθη το ερώτημα, ετέθη πριν από έξι χρόνια από τον ασφαλιστικό τομέα, όπου ε, αναφέρθηκε ότι αν πρόκειται για χρηματοψηφιακά εργαλεία να υπάρχει η σκέψη ότι υπάρχουν ήδη στη μία πλευρά των ισολογισμών θα πρέπει να αναφέρονται και στην άλλη πλευρά των ισολογισμών. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχει κάποια σύγχυση ε, και αυτή την έχουμε διαπιστώσει και στο Διοικητικό Συμβούλιο ε, του ΕΦΡΑΓ όπου καλέσαμε εκπροσώπους να μας πούνε ποιο είναι το πρόβλημα. Και το πρώτο που αναφέρθηκε είναι η μεταβλητότητα ε, στα κέρδη και στις ζημιές. Και αν το λύσουμε αυτό το πρόβλημα θα μπορούσαμε να πούμε ότι λύνεται το πρόβλημα με την κατάργηση της μεταβλητότητας. Το θέμα είναι τώρα το εξής. Η εικόνα είναι ολοκληρωμένη ή μήπως υπάρχουν και άλλα αίτια γιατί είναι προτιμότερο να ακολουθηθεί η άλλη μέθοδος. Νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε έτσι ώστε ο οργανισμός ISB να προσφέρει την εναλλακτική λύση. Αυτό θα γίνει μέχρι μέσα σε δύο εβδομάδες και εκεί θα δούμε ε, κατά πόσο η μία ή η άλλη επιλογή ή και τα δύο σε συνδυασμό θα βοηθήσουν τον ασφαλιστικό τομέα να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Εγώ προσωπικά, όπως και εσείς, ε, θεωρώ ότι είναι πιο λογικό να υπάρξει ε, μετάθεση, χρονική μετάθεση αν σας κατάλαβα καλά, γιατί εμένα, για μένα δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή να ακολουθήσουμε μία ολιστική προσέγγιση. Ο κύριος Άσλεϊ. Ε, συμφωνώ, αλλά το μόνο που ε, δεν θα έλεγα είναι το εξής αν έχει κανείς ε, πέντε ασφαλιστικές εταιρείες μέσα σε μια αίθουσα θα έχει πληθώρα απόψεων για το πώς να λυθούν τα προβλήματα. Αυτά είναι γνωστά και νομίζω όλοι ε, έχουν διαφορετική θέση γιατί ξέρετε κάτι, σε μεγάλο βαθμό ε, πρόκειται για εθνικούς οργανισμούς, έχουν προκύψει από τις εθνικές αγορές και κατ' ουσίαν ε, διαφέρουν στα προϊόντα που προσφέρουν γιατί υπάρχει κάποια ευελιξία. Ε, εγώ λοιπόν ε, πιστεύω ότι η ολιστική προσέγγιση μπορεί να βοηθήσει κάποιους. Δεν θα τα σώμουτα απαραίτητα υπέρ της χρονικής μετάθεσης. Βέβαια δεν μπορούμε να την επιβάλλουμε την ολιστική προσέγγιση ε, γιατί υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και ίσως θα πρέπει κανείς για σύντομο χρονικό διάστημα να δεχτεί αυτές τις διαφορετικές απόψεις. Λέω πρώτα και εγώ είπα ολιστική προσέγγιση ε, για κάποιο χρονικό διάστημα. Πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε. Προφανώς. Δεν είπα ότι είναι τέλεια η fair value, αλλά είναι σημαντικό σε αυτή τη συζήτηση για το fair value και πάλι ζητώ συγγνώμη που κάπως διευρύνω το πεδίο, το πεδίο της συζήτησης. Θα πρέπει λοιπόν να θυμόμαστε ότι πολλές φορές αυτή η συζήτηση για το fair value έχει γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από πλευρά των τραπεζιτών που ήθελαν να ε, παραπλανήσουν το κοινό ε, όσον αφορά τα ε, συσολογισμούς τους. Όταν ε, στις αρχές του 2008 ήταν πολύ έντονη συζήτηση για αυτά τα θέματα με τον κύριο Σάλιβαν που ήταν ο βασικός υποστηρικτής του συστήματος του Fair Value και μάλιστα είδαμε μετά από λίγους μήνες γιατί ασχολήθηκε τόσο με αυτή τη συζήτηση. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να το έχουμε υπόψη μας διαρκώς. Δεν είπα ότι είναι το τέλειο σύστημα γιατί είναι ανοιχτό στην χειραγώγηση αλλά δεν είναι και από μόνο του ε, κακό το σύστημα. Ωραία, έχουμε μια πιο καλή, πιο ξεκάθαρη εικόνα για να τα σκεφτούμε και εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο που είναι όπως ξέρετε ένας φορέας που ακούει ε, και μετά ε, εξετάζει και συζητά τις διάφορες απόψεις. Για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου αναφέρω, ήταν έτσι. Ε, θα το κάνουμε αυτό που είπατε, δηλαδή θα ζητήσουμε τη γνωμοδότησή τους. Να ευχαριστήσω τους ε, ειδικού μας και όλους τους υπόλοιπους για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή συζήτηση. Διακόπτουμε για πέντε λεπτά.